ως διοίκηση σε περιοχές κρίσης είναι κάτι το οποίο απορρίπτουμε. Και με αυτό συμφωνούν και πολλές οργανώσεις της ε, κοινωνίας ε, των ε, πολιτών. Και ακριβώς αναρωτιέμαι πού έλαβε τις πληροφορίες ο συνάδελφος των σοσιαλιστών. Εμείς έχουμε υποβάλει μια σχετική τροπολογία που τα απορρίπτει όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ σας. Ευχαριστώ. Κούκαν, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συζητητές για τη δουλειά που έχουν κάνει εδώ. Όταν είδα την πρόταση της Κομισιόν ε, πρώτη φορά ήμουν πολύ επιφυλακτικός ως πρώην εισηγητής ε, στα σχετικά μέσα. Είδα κάποια προβλήματα στην συγχώνευση όλων των εξωτερικών μέσων υπό μια στέγη. Θα πρέπει λοιπόν να διατηρηθεί η αρχική φιλοσοφία αυτού του μέσους... ένα μέσο το οποίο οδηγεί η πολιτική μας. Και στηρίζοντας την αρχή περισσότερα για περισσότερα, μια αρχή την οποία είχαμε ακριβώς για να ανταμείψουμε τις μεταρρυθμιστικές προτάσεις που οδηγούν σε εδραίωση της δημοκρατίας, κράτους δικαίου και λοιπόν μεταρρυθμίσεων. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δημιουργήσουμε το κατάλληλο πλαίσιο για την ε, συζήτηση της απόδοσης και της κατανομής των σχετικών κονδυλίων. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εμπλακεί περισσότερο στον σχεδιασμό, προγραμματισμό και παρακολούθηση των μέσων αυτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Κώστα έχει το λόγο. Σίλβια Κώστα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και εγώ όλου του συζητητές. Πρέπει να πω ότι ο νέο αυτό μηχανισμό για την εξωτερική πολιτική που περιλαμβάνει και τον μηχανισμό για την πολιτική γειτονία δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε σύγχυση πολιτικών στόχων και διαφορετικών ιδιαιτεροτήτων όσον αφορά την πολιτική, αλλά θα πρέπει να μα βοηθήσει να συνεργαζόμαστε πολύ πιο αποφασιστικά και σε τομείς όπω ο πολιτισμό και η εκπαίδευση. Και βλέπω ότι προωθείται ιδιαίτερα και η πολιτιστική συνεργασία μέσω του μηχανισμού αυτού, κάτι το οποίο εμείς ανέκαθεν λέγαμε ότι θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Για πρώτη φορά στα πλαίσια ενό τέτοιου μηχανισμού διεθνού συνεργασία προβλέπονται κονδύλια τα οποία θα μπορούσαν να δοθούν για να υποστηριχθεί το Erasmus Mundus σε συνεργασία με τρίτε χώρε, πράγμα το οποίο μα είχαν ζητήσει πάρα πολλοί φοιτητέ, μαθητέ από τι χώρε γειτονία ή από την Αφρικανική Ήπειρο. Και επίση χαίρομαι πάρα πολύ που οι εισηγητέ λάβαν υπόψη την πρόταση τη δική μου τη Επιτροπή να ενισχυθούν οι διμερεί διεθνεί σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτε χώρε σε όλε της διμερείς Συμφωνίας και στα πλαίσια της νέας πολιτιστικής ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να προωθήσουμε τον διαπολιτισμικό, διαθρησκευτικό διάλογο και θα καταφέρουμε να, καταφέρουμε, να φέρουμε πιο κοντά όλους εμπλεκόμενους παράγοντες στον τομέα του πολιτισμού. Η κυρία Αντρικέν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στα πλαίσια τη εξωτερική πολιτική χρειαζόμαστε συνέχεια, συνεκτικότητα και συνέπεια και χρειαζόμαστε βέβαια και αποτελεσματικέ εξωτερικέ δράσει και πολιτικά μέσα τα οποία θα έχουν πραγματικά μια σημαντική ε, επιρροή που θα βαρύνουν. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό ο μηχανισμό γειτονία ανάπτυξη διεθνού συνεργασία περιλαμβάνει όλε αυτέ τι διαφορετικέ πτυχέ. Πολλά υπόθηκαν σήμερα από τους εκπροσώπους των τριών αυτών επιτροπών και από τους τέσσερι συνεισηγητές θα ήθελα να σταθώ σε κάποιε πτυχέ. Καταρχά, η χρηματοδότηση από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το μηχανισμό αυτό και όσον αφορά την πολιτική γειτονία πιο συγκεκριμένα. Η πολιτική γειτονία είναι πάρα πολύ σημαντική, εντάσσεται στι συνθήκε μα. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να δοθούν περισσότερα κονδύλια στην πολιτική γειτονία, αλλά δυστυχώ δεν υπάρχει απαραίτητη συμφωνία αυτή τη στιγμή μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την πολιτική γειτονία. Επίσης, Πρέπει να δούμε αν ο μηχανισμός αυτός αντιστοιχεί στις ε, φιλοδοξίες μας για την ε, προστασία του ε, πολυμερού συστήματος εμπορίου. Και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπενιφέ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόταση συγχώνευσης των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης όσον αφορά την ανάπτυξη, την πολιτική γειτονίας, την αναπτυξιακή συνεργασία, μολονότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποιε ανησυχίε. Θεωρώ ότι η επέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν ιδιαίτερα καθοριστική προκειμένου να διασκεδαστούν οι ανησυχίε αυτέ. Και χαίρομαι που βλέπω ότι έχουν ενσωματωθεί οι προτεραιότητε Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων όσον αφορά τα μέσα εξωτερική χρηματοδότηση, όσον αφορά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσον αφορά την δημοκρατική λογοδοσία. Ο ρόλο του ενισχύεται. Επίση, απλουστεύεται το όλο σύστημα και αυτό είναι σημαντικό. Η πολιτική γειτονία θα πρέπει να έχει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο και να προβλέπεται αρεσιμότητα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου μόνο αν τηρούνται οι προποθέσει αυτέ να χρηματοδοτούνται μέσω των μέσων αυτών τρίτε χώρε. Θα πρέπει η πολιτική μα να είναι αξιόπιστη και θα πρέπει πραγματικά να καταφέρουμε να προωθούμε θεμελιώδεις αρχές και αξίες ακόμη και όταν προωθούμε ευρωπαϊκές, ευρωπαϊκά ή εθνικά συμφέροντα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε μια πολιτική γειτονία που θα προωθεί την ειρήνη και να στραφούμε κατά οποιασδήποτε απόπειρα επικιοκρατία που έρχεται από οποιαδήποτε πλευρά. Ο κύριος για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Επίτροπε, Αγαπητή Επίτροπε, μάλλον κύριε, ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι πολύ χρήσιμος αυτός ο μηχανισμός και εδώ και πολύ καιρό μας βοηθά να προωθήσουμε τις αρχές και αξίες μας. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να συνενώσουμε τα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης και να προβλέψουμε ελαστικότητα ε, σε ό,τι αφορά τη χορήγηση αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά όχι ει βάρο ε, της δημοκρατίας και των μηχανισμών ελέγχου. Συμφωνώ με τις τροπολογίες πρέντα εκ μέρους του ΕΛΚ που ζητούν ένα ξεχωριστό μέσο για την πολιτική γειτονία και επίση τονίζουν την πολιτική σημασία που έχουν οι σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τι γειτονικέ της χώρε. Θα πρέπει ιδιαίτερη προσοχή να αφιερώσουμε στην πολιτική γειτονία μα και επίση να την αντιμετωπίσουμε ξεχωριστά και να μην την εντάξουμε στη γενική αναπτυξιακή πολιτική μας. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Ενρίκε Γκερέρο Σαλόμ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αν χρησιμοποιήσουμε επαρκώς, αλλά μόνο αν χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα αυτό το μηχανισμό, μπορεί να αποτελέσει μηχανισμό που θα κάνει πιο συνεκτική τη φωνή και πιο ε, στεντόρια τη φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο εξωτερικό και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη φωνή για να προωθούμε δημοκρατικές αξίες, ε, κοινωνική βιωσιμότητα, προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεργασία, ειρήνη και σταθερότητα. Μόνο έτσι θα χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα αυτό το μηχανισμό. Και ως ηγητής ανθρωπιστικής βοήθειας εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαπίστωσα κατά τη διάρκεια των συζητήσεων πώς έχουν αλλάξει φύση οι ανθρωπιστικές κρίσεις γιατί οι μεμονωμένες κρίσεις έχουν ε, μετατραπεί σε ε, μακροχρόνιες κρίσεις και χρειάζεται άμεση ε, ενίσχυση για την αντιμετώπιση των αναγκών. Αν χρησιμοποιήσουμε λοιπόν το μηχανισμό αυτό για να διαφυλάξουμε την ειρήνη ή να την ανασυγκροτήσουμε όταν παραβιάζεται, τότε θα αξίζει πραγματικά ο μηχανισμός αυτός την υποστήριξή μας στην αυριανή ψηφοφορία. Σας ευχαριστούμε κύριε Γκερέρο Σαλόμ. Το λόγο έχει ο κύριος ε, Μπογδάν Σδρογεύσκη. Από... Σας ευχαριστώ. Από τα μέχρι τώρα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης και της εξωτερικής δράσης ε, λήγουν στα τέλη του επόμενου χρόνου. Ε, γι' αυτό θα πρέπει να τα αντικαταστήσουμε και χαίρομαι με τη διόρθωση και τις αλλαγές που προτείνονται. Γιατί αξιοποιούμε τις εμπειρίες μας, καλές και κακές, για να βελτιώσουμε τις ε, επιδόσεις μας. Και δεν μιλάμε για ε, αμεληταία κονδύλια, μιλάμε σχεδόν για 90 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε με τα κονδύλια αυτά την, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα αποτελεσματικής, αποτελεσματικής δράσης υπέρ της δημοκρατίας και των άλλων αξιών που προσπίζουμε. Εκ μέρους της Επιτροπής Πολιτισμού θα ήθελα να απευθύνω έκκληση να χρησιμοποιήσουμε ε, κάποιους μηχανισμούς όπως το Erasmus Plus, η Δημιουργική Ευρώπη ή το Ορίζοντα 2020 που ολοκληρώνεται και που είναι συναφή προγράμματα να ε, αξιοποιήσουμε τις εμπειρίες από όλα αυτά τα εκπαιδευτικά πολιτιστικά προγράμματα και τα προγράμματα ε, ε, υποτροφιών για να εξασφαλίσουμε στο νέο μηχανισμό μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Σας ευχαριστώ. Κυρία Νίνα Γκίλ, έχει το λόγο. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, Επίτροπη. Ο αυξανόμενο αριθμός των παγκοσμίων προκλήσεων σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματική. Βεβαίω είναι ένα θέμα αυτό, αλλά πρέπει να εστιάσουν πολύ περισσότερο στην πολιτική και τον συντονισμό των προγραμμάτων με τα κράτη-μέλη βλέπω πως ε, η πρόταση της ε, Κομισιόν ε, ελπίζω μάλλον να συμβαδίσει με μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Η ερώτησή μου είναι πρώτα απ' όλα εάν θα συμφωνήσει η Κομισιόν σε κάποια κριτήρια για αναστολή χρηματοδότησης σε χώρες που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεύτερον, η έκθεση αυτή προτείνει μια καλύτερη ευθυγράμμιση των χρηματοδοτήσεων αυτών με τους στόχους των Παρισίων. Θα δεσμευτεί η Κομισιόν για τους στόχους αυτούς τρίτων. Έχουμε εδώ πέρα ένα πλαφόν στην βοήθεια που θα πάει σε στρατιωτικές ε, δραστηριότητες ε, ακριβώς για να βοηθήσουμε στην ανοικοδόμηση και όχι στην άμυνα. Ελπίζω να ισχύσει αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Γκίλ. Κυρία Ζέλιανα Ζόφκο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, συνοπητοί συνάδελφοι. Ε, βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει πρόβλημα με την ενότητά μας. Μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις με μια ενιαία προσέγγιση στην εξωτερική δράση και στενότερη αναπτυξιακή συνεργασία. Πρέπει να μεγιστοποιήσουμε την προσθέμενη αξία και να μοιραστούμε τις εμπειρίες όλων των κρατών μελών μαζί. Θα μπορέσουμε να επιτύχουμε πολύ περισσότερα από κάθε κράτος μέλος μόνο του. Για να επιτύχουμε αυτούς τους ε, στόχους εγώ μαζί με τους άλλους συναδέλφους ε, που συνυπογράφουμε υποβάλαμε την ε, τροπολογία υπαριθμών 555 που ζητάει να αυξήσουμε τη συνεργασία και τις ικανότητες μας αγαπητοί συνάδελφοι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας και στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για να προωθήσουμε ακριβώς ε, τα μέσα αυτά και να μπορέσουμε να δράσουμε από κοινού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφε. Και τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Κιέγγε για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Η εξάλληψη της ε, φτώχεια είναι ο πρωταρχικό στόχο τη αναπτυξιακή συνεργασία. Η εξωτερική δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμπορεύεται με τι μεγάλε παγκόσμιε προκλήσει, ιδιαίτερα με την επίτευξη των στόχων τη Ατζέντα 2030. Με την έγκριση του Μηχανισμού Γειτονία, Ανάπτυξη και Διεθνού Συνεργασία, κάνουμε ένα ακόμα θετικό βήμα για την καταπολέμηση τη ένδυα, Είτε πρόκειται για οικονομική, δημοκρατική, κοινωνική ή περιβαλλοντική ένδια. Ο νέος και φιλόδοξος αυτός μηχανισμός θα δώσει τη δυνατότητα να έχουμε μια μεγαλύτερη ισχύ, να μπορούμε να επέμβουμε μεγαλύτερη ισχύ όσον αφορά τις οικονομικές αξίες της δημοκρατία, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικονομικής ενσωμάτωσης, καθώς επίσης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Πρέπει να τονίσω ότι η νέο μέσο δεν σημαίνει έλλειψη διαφοροποίησης. Το αντίθετο, μάλιστα, οι γραφικέ προτεραιότητε θα συνεχίσουν να έχουν πολύ μεγάλη σημασία, όπω για παράδειγμα για τι νέε συμφωνίε με τι χώρε ΑΚΕ. Η καινοτόμα και νέα φύση του νέου αυτού μηχανισμού θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βαρύνει ακόμα περισσότερο στο διεθνέ προσκήνιο, όπου μόνο μια συνεκτική και ολιστική προσέγγιση θα είναι αποτελεσματική. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Περνάμε τώρα στην διαδικασία και Eye. Μπορώ να δώσω τον λόγο σε όλους τους ε, συναδέλφους. Η κυρία Σόιντροβα πρώτη για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Παρακολούθησα την συζήτηση πολύ προσεκτικά και μας δείχνει ότι δεν υπάρχει κάποια ενότητα για το τι μορφή πρέπει να έχει αυτό το μέσο. Και παρόλα αυτά είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο και για τις ε, χώρες αυτές ε, και για τις χώρες της ε, γειτονία. Ένα πάρα πολύ μεγάλο μέσο μπορεί να αλλάξει την πραγματικότητα στις χώρες αυτές και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη αυτών των χωρών. Μπορούμε να προλάβουμε άλλες μεταναστευτικές κρίσεις Οπότε έχει τεράστια σημασία να το προετοιμάσουμε σωστά. Αντιλαμβάνομαι πως η Κομισιόν θέλει να το κάνει πιο αποτελεσματικό, να συγχωνεύσει διάφορα μέσα σε ένα, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με τρόπο λογικό και διαφανή για τους δικαιούχους σύμφωνα με τις ΜΚΟ ε, φοβούνται την ε, απώλεια της στήριξης που έχουν αυτή την στιγμή. Γι' αυτό στηρίζω το αίτημά τους για το πρόγραμμα για την πολιτική γειτονία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Julie Ward τώρα για ένα λεπτό. Στην εποχή του Τραμπ και του Μπολσονάρο και των πρακτόρων του Πούτιν που αναμειγνύονται στις δημοκρατικές διαδικασίες, η διεθνή συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντική. Χαίρομαι που βλέπω πως περιλαμβάνονται οι συστάσεις της Επιτροπής Πολιτισμού στο κείμενο. Παραδείγματος χάρη, το Κοινοβούλιο στηρίζει την χρήση αυτού του μέσου για τα προγράμματα Creative Europe και Erasmus Plus. Έτσι θα ενισχυθεί σημαντικά η πολιτιστική διάσταση και η πολιτιστική διπλωματία μέσω των άμεσων επαφών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να υπάρχει μια αλληλοκατανόηση και εμπιστοσύνη και να ενισχυθεί η δημοκρατική ζωή. Σε έθραστες δημοκρατίες και χώρες που βγαίνουν από συγκρούσεις Συχνά ο πολιτισμός και ο αθλητισμός δημιουργούν την βάση ανοικοδόμησης κοινωνιών. Σας ευχαριστούμε κυρία Γουόρντ. Τώρα θα δώσω τον λόγο στον Ζόρντι Σουλά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι με το νέο μηχανισμό γειτονίας ανάπτυξης και τεθνούς συνεργασίας τα χρήματα ε, και τα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης θα πλουστευθούν και έχουμε μεγαλύτερη κατανόμη των κονδυλίων και περισσότερα κονδύλια, κάτι που θα ενισχύσει τις εξωτερικές δράσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως ε, θα πρέπει να επικεντρωθούμε κυρίως στο εξή ερώτημα. Ο νέος αυτός μηχανισμός θα εξυπηρετήσει κυρίως ε, το στό, τους γεωπολιτικούς στόχους και τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μήπως θα προωθήσει κυρίως την επίτευξη των διεθνώς αναγνωρισμένων αρχών της αναπτυξιακής βοήθειας και της διεθνούς συνεργασίας. Με άλλα λόγια, το, ο νέος μηχανισμός γειτονίας Ανάπτυξη και διεθνούς συνεργασίας θα καταστήσει ε, τη ε, χορήξη αναπτυξιακής βοήθειας όμοιρο ε, των πολιτικών ελέγχων της μετανάστευσης θα χρησιμοποιήσει για την πρόσπιση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ειρήνης, της πρόληψης ε, των συγκρούσεων και της προστασία του περιβάλλοντος, θα πρέπει να φροντίσουμε οι φιλοδοξίες και οι στόχοι του νέου μηχανισμού να είναι η σωστή και κατάλληλη για το νέο πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σόλε. Ο κύριος Πόλτσακ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η πολιτική γειτονία και η αναπτυξιακή πολιτική είναι ταυτόχρονα και μέσα εξασφάλιση ε, τη ε, ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μα ενδιαφέρει όχι μόνο η εσωτερική αλλά και η εξωτερική μα ασφάλεια. Και γι' αυτό χαιρετίζω ε, τη πρικοδότηση του νέου μηχανισμού από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Επίσης, με τη συγχώνευση των προηγούμενων προγραμμάτων σε ένα νέο πρόγραμμα θα ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα των δράσεών μας και θα αξιοποιήσουμε καλύτερα τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Κάθε Πέμπτη συζητούμε στην Ολομέλεια την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο και με τη δημιουργία της πολιτικής αιρεσιμότητας και την επιμονή μας στις δημοκρατικές αρχές θα προωθήσουμε τις αξίες μας και θα βελτιώσουμε τον αντικτύπο των πολιτικών μας. Ευχαριστώ. Ο λόγος και πάλι στον Επίτροπο, τον κύριο Μίμητσα. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω κάποιες ερωτήσεις που έγιναν απευθείας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω αν ε, θα τις απαντήσετε, γιατί ε, ρωτήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι θα γίνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα, αν ο μηχανισμός θα συμπεριλάβει και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι η ευκαιρία σας τώρα να απαντήσετε σε όλες αυτές τις απορίες των Ευρωβουλευτών. Ε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Σας ευχαριστώ για την πολύ χρήσιμη αυτή συζήτηση που είχαμε και να σας χαρώ ακόμη μια φορά για την αποφασιστικότητα που δείξατε για να καταλήξετε στην ολοκληρώστε μάλλον την πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τόσο εγκαίρος. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις όταν θα είναι έτοιμο και το Συμβούλιο. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ομόφωνα Είμαστε πεπισμένοι ότι το να δημιουργήσουμε έναν συνεκτικό και πιο υπεύθυνο μηχανισμό αναπτυξιακή βοήθειας αποτελεί πραγματικά ένα πολύ θετικό βήμα για να πετύχουμε του στόχους μας και να τηρήσουμε τις δεσμεύσει μας στο πλαίσιο της παγκόσμια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της, συνένωσης, Ευρωπαϊκή συνένεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη στα πλαίσια της Ατζέντα 2030. Και τονίζω και επαυξάνω ότι ε, όλα αυτά θα βασιστούν στην αρτεκτονική την οποία εγκρίνεται στα πλαίσια της έκθεσης αυτής μέσω συγκεκριμένων μέτρων, δίνοντας πολιτική σημασία σε κάθε θεματική, γεωγραφική πολιτική, συμπεριλαμβανομένως βέβαια και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Κατά την άποψή μας, οποιαδήποτε τροποποίηση που θα μπορούσε πραγματικά να υπονομεύσει τη συνεκτική αυτή δομή του μηχανισμού αυτού, όπως υποστηρίζεται από την έκθεση αυτή, ουσιαστικά θα οδηγήσει σε ασυνέπεια και σε πολλές αντιφάσεις μεταξύ των πολιτικών μας στόχων και, των, και της ικανότητας χρηματοδότησης των στόχων αυτών και της ικανότητας χρηματοδότησης των πολιτικών μας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό είμαι πεπισμένος ότι ε, το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια ξεχωριστά μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης ουσιαστικά δεν δίνουν ιδιαίτερη αξία σε κάποια συγκεκριμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έλεγα το αντίθετο μάλιστα, ότι ε, το καλύτερο είναι να καταφέρουμε να έχουμε μια γενικότερη σφαιρική πολιτική και μια καλύτερη συνεκτικότητα όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε. Αυτό όσον αφορά και τους εξωτερικούς μας εταίρους. Και θα ήθελα επίση να επιστήσω την προσοχή σας, αξιότιμα μέλη, στο ότι ε, τα μέσα χρηματοδότησης τα οποία προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις ε, προτεραιότητες που έχουμε στα πλαίσια της αναπτυξιακής βοήθειας όπως οι προτεραιότητες αυτές καθορίζονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Συνένεσης για την Ανάπτυξη. Επομένως, τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν μια κέρια βάση, θα πρέπει να εξαλείψουμε σε κάθε περίπτωση την φτώχεια, θα πρέπει να έχουμε μια δημοκρατική προσέγγιση βάσει συγκεκριμένων κανόνων για όλους τους εταίρους μας. Όλα αυτά αποτελούν σταθερές μας αξίες και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακολουθούμε μια συγκεκριμένη πολιτική εφαρμογή και μια παρακολούθηση τη σωστή εφαρμογή όλων αυτών των χρηματοδοτικών μέσων. Τώρα, όσον αφορά όλου αυτού του συναδέλφου, οι οποίοι εξέφρασαν κάποιε ανησυχίε, όσον αφορά το ενδεχομένω να παρεκκλίνουμε από και να κινηθούμε περισσότερο προς τη χρηματοδότηση αμυντικών ή στρατιωτικών στόχων. Προς αυτούς λοιπόν τους συναδέλφους θα έλεγα το εξής. Αν δούμε τις ε, βασικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, θα συνειδητοποιήσετε ότι οποιαδήποτε αμυντική δράση που χρηματοδοτείται, που θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τον κοινωτικό προπολογισμό, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί ουσιαστικά στην πράξη. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο και αυτό θα συνεχίσει να αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο τη πολιτική που θα ακολουθήσουμε και στο μέλλον για την ανάπτυξη. Για ακόμη μια φορά να τονίσω το εξή οι στόχοι που έχουμε στα πλαίσια της επιλεξιμότητας των κονδυλίων για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια ακολουθούν μια απόλυτη ισορροπία σε σχέση με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να έχουμε μια καλύτερη κατανομή των κονδυλίων αναγεωγραφική περιοχή ή ανα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προβλέπεται εδώ και απαραίτητη ευελιξία. Για ακόμη μια φορά θα ήθελα να επιβεβαιώσω τη δέσμευσή μας για ένα ανοιχτό διάλογο με εσά, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια δίκαιη και ισορροπημένη λύση, προκειμένου να καταφέρουμε να ενισχύσουμε τον εποπτικό ρόλο ή τον πολιτικά καθοδηγητικό ρόλο που θα μπορούσε να λάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για μια ακόμη φορά λοιπόν σας ευχαριστώ και προσβλέπω σε μια θετική δική σας ψήφο αύριο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Και τώρα θα ξαναδώσω το λόγο στους συνεισηγητές, που είναι τέσσερις, ξεκινώντας από τον κύριο Αντώνιο Παντσέρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα το αν μπορούμε να έχουμε μια ικανότητα σφαιρικής αντιμετώπισης των προτεραιοτήτων μας και αν καταφέρνουμε από την άλλη να συνδυάσουμε το σφαιρικό αυτό όραμα με συγκεκριμένους τοπικούς, πολιτικούς, γεωγραφικούς στόχους. Με αυτή ακριβώς είναι η ισορροπία που προσπαθήσαμε να πετύχουμε και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο ορισμένοι συνάδελφοι ανησυχούν αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κανένα λόγο ανησυχία που να απορρέει από τον νέο αυτό μηχανισμό γειτονία, ανάπτυξη και διεθνού συνεργασία. Τους τελευταίους αυτούς μήνες υπήρχαν πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι ήταν τόσο υποστηρικτές, θα έλεγα, ένθερμοι θειασότες της πολιτικής γειτονίας και είναι αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι ήταν έτοιμοι να θυσιάσουν την πολιτική αυτή στο όνομα άλλων πολιτικών. Η πολιτική αυτή πλέον ενσωματώνεται στον νέο αυτό μηχανισμό. Η διακυβέρνηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το τονίζω, εμπλέκεται όλο και περισσότερο, ελέγχει όλο και περισσότερο μέσω κατεξοδότηση πράξεων και μπορεί κατά αυτόν τον τρόπο στα πλαίσια του προγραμματισμού να καθορίζει τι βασικέ πολιτικέ στρατηγικέ που θα ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα τη ανάπτυξη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δυστυχώ κανεί δεν τον έφερε αυτό το πράγμα. Θα έχουμε ένα υψηλότερο βαθμό διαφάνεια και μπορεί πλέον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το μηχανισμό αυτό να συναποφασίζει στην ουσία. Τρίτον, νομίζω ότι είναι υπερβολικό αυτό που κάποιοι συνάδελφοι που είπαν ότι ο μηχανισμό αυτό ουσιαστικά δημιουργήθηκε για να αναχαιτιστεί η μετανάστευση. Ας μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές αυτές οι μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις μας κάνουν να μην βλέπουμε τελικά τη μεγάλη αξία που έχει ένα τέτοιο μηχανισμό, ο οποίο μπορεί να προωθήσει πραγματικέ σφαιρικέ πολιτικέ τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα τη αναπτυξιακή συνεργασία. Τέλο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Πρόεδρε, να καταφέρουμε μέσω του μηχανισμού αυτού να πετύχουμε ένα σημαντικό ποιοτικό άλμα για την εξωτερική πολιτική αλλά και την πολιτική αναπτυξιακή συνεργασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, καταδεικνύοντα πραγματικά ότι μπορούμε να προωθούμε πολιτικέ συνεκτικέ και να καταφέρουμε ουσιαστικά να καλύψουμε όλα αυτά τα κενά τα οποία είχαμε τα τελευταία χρόνια. Σας ευχαριστούμε, Σας ευχαριστούμε κύριε Παντσέρη. Περνάμε τώρα στον συγητή από την Επιτροπή Εξωτερικών, τον κύριο Πρέντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να διευκρινίσω την τροπολογία που κατέθεσε εκ μέρους του ΕΛΚ ε, και που αφορά το ψήφισμα που συνοδεύει την έκθεση. Ε, που δεν είναι στόχος μου να ματαιώσω τις προσπάθειες και τα κοινά επιτέγματα των τελευταίων 8 μηνών. Και όντω καταφέραμε να βελτιώσουμε τα πράγματα για τη γειτονία. Αυξήσαμε κατά 24% τα κονδύλια της γειτονία. Επίσης ενισχύσαμε το πολιτικό πλαίσιο της γειτονία που είναι βασικό τομέα τη εξωτερική μας δράσης. Επίσης βελτιώσαμε την προσέγγιση που στηρίζεται πια στις επιδόσεις, τα αποτελέσματα. Ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής πολιτικής της γειτονία. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να δείξουμε ρεαλισμό και να πούμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Η λύση ακόμη... Ε, ενός ξεχωριστού μηχανισμού γειτονίας παραμένει στο τραπέζι ανοιχτή. Το Συμβούλιο εξακολουθεί, να είναι διχασμένο για τα θέματα γειτονία. Οπότε θα πρέπει να αφήσουμε όλες τις δυνατότητες ανοιχτές για το επόμενο ε, κοινοβούλιο που θα ξεκινήσει τη διαπραγματεύση. Γιατί μας αρέσει είτε όχι, προς το παρόν ο Μηχανισμός Γειτονίας Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας είναι ένας γίγαντας με πόδια. Επίσης, ε, στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, όπω είπε και ο κύριος Παντσέρη, ε, υπήρξε ε, ο πειρασμός από τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης να ε, οικειοποιηθούν τον όλο μηχανισμό ακολουθώντας μόνο το πρίσμα της ανάπτυξης και ε, ε, να βγάλουμε τις χώρες της Βόρειας από την νότια γειτονία και να, καλέσουμε μόνο, να κρατήσουμε μόνο τις χώρες μέσα της Ανατολής ε, στη γειτονία και τις χώρες της Ανατολής. Όχι, είναι απαράδεκτο να διαταράξουμε αυτή την πολιτική μόνο και μόνο για ένα μηχανισμό, ούτε να θέλουμε να μονοπολίσουμε τη διεθνή συνεργασία μειώνοντας την εξωτερική πολιτική μας και την ε, πολιτική γειτονία μας. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να θετούμε μια πολιτική προσέγγιση. Οι γείτονέ μας είναι πολύ πιο σημαντικοί από οποιοδήποτε άλλο σε ό,τι αφορά τα χρηματοδοτικά μας μέσα. Δεν μπορούμε να το αγνώμουμε αυτό, ούτε να θυσιάζουμε τις γειτονικέ μας χώρες στο όνομα ενός αφηρημένου συμφέροντος και για να εξασφαλίσουμε περισσότερα κονδύλια, για να τροφοδοτούμε ε, ουτοπικά όνειρα. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρέντα. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Φρανκ Έγκελ, ο εισηγητής της Επιτροπής Ανάπτυξης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. δεν θα το πάρω προσωπικά, παρόλο που θα μπορούσα αυτό που είπε ο κύριος Πρέντα. Ακούσαμε πολλές ανοησίες από την άκρα αριστερά σήμερα. Ε, που χρειάστηκε να τις ε, χωνέψουμε εδώ και πολλούς μήνες, ότι είναι μιλιταριστικό στρατιωτικο, ε, ε, όργανο στρατιωτικοποίησης και ούτω καθεξής. Κι όμως ο μηχανισμός αυτός είναι ενδιαφέρον και θα μας επιτρέψει να εφαρμόσουμε τη στρατηγική μας για την Αφρική, που ζητούμε σε κάθε διάσκεψη κορυφής τα τελευταία δύο-τρία χρόνια και μέχρι στιγμής λόγω έλλειψης ε, συνεκτικής χρηματοδότησης δεν, κατάφερα, δεν καταφέραμε να υλοποιήσουμε. Επίσης, ε, θα έχουμε καλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ των εδαφών που καλύπτονται από την πολιτική γειτονία και των εδαφών που καλύπτονται από την πολιτική συνεργασία. Κάτι που έχει νόημα, γιατί δεν μπορούμε τη σήμερα ημέρα να ε, ξεχωρίζουμε την Αλγερία από τον Ήγηρα, τη Λιβύη από το Τσάντι, το Μαρόκο από τη Μαυριτανία. Υπάρχει στενή αλληλεπίδραση μεταξύ των χωρών που καλύπτονται από τη μία πολιτική και των χωρών που καλύπτονται από την άλλη πολιτική. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένε οι χώρε και γι' αυτό έχει νόημα ο ενίο μηχανισμό. Επίση, διαφυλάσσουμε ανοιχτέ όλε τι δυνατότητε για τη συνέχιση τη εταιρική σχέση με τι χώρε ΑΚΕ. Είναι σημαντικό από του χρόνου που θα αντικατασταθούν οι συμφωνίε του Κοτών από κάτι άλλο, που δεν ξέρουμε τι ακριβώ θα είναι. Είναι σημαντικό όμω στο μέλλον ο νέος μηχανισμός να καλύπτει όλες τις πιθανότητες. Γενικώ πιστεύω ότι ο νέος μηχανισμός είναι θετικός γιατί περιλαμβάνει και τη γειτονία μεταξύ άλλων. Και μακάρι αύριο να εγκρίνουμε αυτή την έκθεση και να παραμείνει ο μηχανισμός με τη μορφή που έχει. γιατί μερικές φορές υπάρχει και φετιχισμός και όχι μόνο πολιτικός ρεαλισμός. Θα πρέπει να έχουμε σε συνεπή και φιλόδοξη χρηματοδότηση όλων των εξωτερικών μας δράσεων. Αυτά σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Γκέρενς, ο τελευταίος μας εισηγητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει για ακόμη μια φορά να επιβεβαιώσω ότι σε συνεργασία με τους υπόλοιπους συνεισηγητές συζητήσαμε απόλυτη ειλικρίνεια, εντελώς ανοιχτά, ανταλλάξαμε επιχειρήματα και αυτό το οποίο μετράει τελικά είναι ο τελικός συμβασμός. Τώρα να προσάπτουμε στον ένα στον άλλον ότι προώθησε τα δικά του επιχειρήματα δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει μόνο το αποτέλεσμα θεωρώ και καταφέραμε να καταλήξουμε στο αποτέλεσμα αυτό με πνεύμα εντελώ επικοδομητικό. Εγώ αυτό κρατάω από την όλη συνεργασία που είχαμε. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, άκουσα τώρα ορισμένου συναδέλφου να λένε πράγματα και ουσιαστικά οι συνάδελφοι αυτοί μάλλον δεν έχουν διαβάσει την έκθεση. Εγώ διάβασα και την ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνέβαλα στην κατάρτιση τη έκθεση αυτή και ορισμένε από τι παρατηρήσει που άκουσα δεν είναι καθόλου δικαιολογημένε. Σε καμία περίπτωση δεν προωθείται εδώ πέρα μόνο η ανάπτυξη. Ένα 95% του μηχανισμού αυτού σαφώς πηγαίνει στην ανάπτυξη. Και ακόμα και η πολιτική γειτονία δίνει τα περισσότερα κονδύλια για την ανάπτυξη. Επομένως, ε, δεν θα πρέπει να έρχονται μερικοί εδώ πέρα να λένε ότι δεν είναι ο μηχανισμός αυτός, ένας μηχανισμός ανάπτυξης. Έχουμε επίσης και διασφάλιση των γεωγραφικών πυλώνων, άρα δεν τροποποιείται τίποτα σε σχέση με την προηγούμενη πολιτική. Αλλάζουμε απλώς μέθοδο αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα κοινό ταμείο, ένα κοινό αποθεματικό για όλους αυτούς τους πυλώνες, για όλα αυτά τα μέσα τα οποία συγχωνεύονται. Και κατά αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Και αυξήσαμε και τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα, ορισμένοι μας δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει ακόμα περισσότερα πράγματα για την αναπτυξιακή συνεργασία. Ως προς αυτό το ακόλουθο. Όχι μόνο κάναμε το μέγιστο, αλλά προσπαθήσαμε να υπερβούμε και τα δυνατά. Και αν είχαμε δώσει ακόμα περισσότερα κονδύλια για την, πολιτική, για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα πρέπει να είχαμε απευθυνθεί στα κράτη-μέλη περισσότερο, που είχαν πει ότι ένα 0,7% θα δινόταν στην επίσημη επιτυξιακή βοήθεια. Αν τα κράτη-μέλη είχαν πραγματικά τηρήσει τις υποσχέσει τους και αν όντω είχαν συνεργαστεί στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε στην περίπτωση αυτή θα μπορούσαμε πραγματικά να δώσουμε στην επόμενη προγραμματική περίοδο τουλάχιστον επιπλέον 200 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Ανάπτυξη. Άρα δεν νομίζω ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή να κατηγορούμε τις Βρυξέλλες στο Στρασβούργο. Θα πρέπει να πάμε στη Ρώμη, στη Μαδρίτη, στη Βαρσουβία, στο Παρίσι, σε όλες τις πρωτεύουσες εκείνες όπου οι κυβερνήσεις δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους. Αν πραγματικά λοιπόν θέλουμε να κάνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση έναν παράγοντα ανάπτυξης, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι μόνο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο. Και λοιπόν που πρέπει να υπενθυμίσω βέβαια όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία είναι προφανή. Θεωρώ λοιπόν ότι η εργασία που επιτελέσαμε μας επιτρέπει να μας επέτρεψε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα στα πλαίσια των τρεμερών διαλόγων με το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο δυστυχώς όμως δεν έχει εργαστεί ακόμα όσο εμεί περιμέναμε. Ελπίζουμε ότι θα σημειώσει πρόοδο στη στάση του και ότι τελικά δεν θα αποκλίνουν πάρα πολλοί απόψει μα με το Συμβούλιο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκέρενς. Ολοκληρώσαμε την συζήτηση. Θα ψηφίσουμε για την έκθεση αυτή αύριο. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Έκθεση του κυρία Σαλαφράγκα Σαντζεσενέρα και έκθεση του κύριου Φλέγγενστάιν όσον αφορά το μηχανισμό προταξιακής βοήθειας, IPA 3. Θα ήθελα να δώσω ευθύ αμέσω το λόγο στους εισηγητές, ο κύριος Σαλαφράγκα πρώτος για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα τον συνεισηγητή μου, τον κύριο Φλέκενστάιν, για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Και θεωρώ ότι αυτή η αγαστή συνεργασία θα μπορούσε να ε, εκλειθεί ως υπόδειγμα καλή συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παράδειγμα προς μίμηση. Επίσης να ευχαριστήσω και τους και οδησηγητές. Κύριε Επίτροπε, πριν να σας κάνω μια σύντομη εισαγωγή στα βασικά στοιχεία της έκθεσης, να σας εκφράσω μία ανησυχία που την εστερνίζονται κάποιοι συνάδελφοι και στα πλαίσια της προεκλογικής φάσης που βρισκόμαστε σε σχέση με τον, τον τίτλο που έχει αυτό το όργανο, ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας 3, ό,τι αφορά τους δικαιούχους του. Ε, και θα πρέπει να διασκεδαστούν στο μέλλον αυτές οι αμφιβολίες για το ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι τελικά του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας. Αυτό ε, τόνισε και πολλοί συνάδελφοι. Επίσης είναι σημαντικό το κονδύλιο αυτού του, του μέσου, περίπου 15 δισεκατομμύρια, πολύ σημαντικό ποσό που θα στηρίξει τις πολιτικές, διοικητικές, οικονομικές, νομικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν στις χώρες που βρίσκονται σε προενταξιακή φάση. Ε, επίσης, ε, αυτά τα μέσα, κυρία Πρόεδρε, ε, ευθυγραμμίζονται και με την ανάγκη ε, τη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της ε, χρηστή διακυβέρνηση και αφορούν και κάποιους συγκεκριμένους τομείς αρμοδιοτήτων που διέπονται από τις αρχές που εμπνέουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανθρώπινα δικαιώματα, θεμελιώδεις ευκαιρίες, κράτος δικαίου και ασφάλεια δικαίου. Επίσης, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, αγροτική ανάπτυξη, γεωργία, έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, ανακτυξιακή πολιτική, προστασία του περιβάλλοντος, καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και κυρίως ε, διαπεριφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία είναι σημαντικά στοιχεία που στηρίζονται, που στηρίζονται από το νέο μηχανισμό. Μία διαφορά του τρίτου ε, μηχανισμού προταξιακής βοήθειας είναι η ακριβωδή κατανομή και η άμεση και έμεση διαχείριση, καθώς και η ανάγκη εμβάθυνσης ε, και της ενίσχυσης της προβολής ε, της χρηματοοικονομικής υποστήριξης Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις χώρες που βρίσκονται σε προεταξιακή φάση. Επίσης, τονίζουμε Τη εξουσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό το μέσο που είναι ε, στα, όπως και ο μηχανισμός ε, γειτονίας Ανάπτυξη και διεθνή συνεργασία, στόχο έχει να ενισχύσει τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μαζί με το Συμβούλιο θα προσδιορίζεται ετήσια κονδύλια στα πλαίσια του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις απόψεις και τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παρακολουθεί όλες τις συζητήσει για τον προγραμματισμό προγραμματισμό και μέσω των κατεξοδότηση πράξεων θα διαδραματίζει ενεργό ρόλο ώστε να έχουμε ουσιαστικό στρατηγικό διάλογο όπου και τα τρία θεσμικά όργανα θα παίζουν τον αντίστοιχό τους ρόλο. Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο και με αυτό θα ολοκληρώσω κυρία Πρόεδρε είναι ότι βρήκαμε έναν ισορροπημένο τρόπο για να συνδυάσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης ε, στην ανάπτυξη όλων των ε, δράσεων του χρηματοδοτικού μέσου και ελπίζω, ε, κύριε Επίτροπε, ότι θα συνεχίσουμε την στενή συνεργασία ώστε να καταστεί αυτός ο μηχανισμός πολύ σημαντικό στοιχείο των υποψηφίων για ένταξη χωρών και της βοήθειας που τους προσφέρουμε. Ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Φλεκεστάιν και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας σε αυτό το ε, θεσμικό τρίγωνο για να υλοποιήσουμε το μηχανισμό πρωταξιακής βοήθειας που είναι απαραίτητο στοιχείο των εξωτερικών μας δράσεων. Ευχαριστώ κύριε Σαλαφράγκα. Το λόγο έχει ο συνεισηγητής, ο κύριος Φλέκενστάιν. Κύρια Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Σάλα για τα καλά του λόγια Έχετε δίκιο ε, για τα όσα είπατε και θα ήθελα να σας τα ανταποδώσω. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και το βασικότερο, ένα θετικό αποτέλεσμα. Το ΜΠΒ3 είναι ένα μέσο ε, το οποίο με 15 εκατομμύρια ευρώ βεβαίως ε, σημαίνει ότι δεν είναι μια τυχαία γειτονία, μιλάμε για μελλοντικά κράτη-μέλη, δηλαδή συγκεκριμένα οι έξι των Βαλκανίων. Το προηγούμενο το Κυριακό ε, είχαμε την επέτειο του βομβαρδισμού του καθιστώτος Μιλόσεβιτς ε, από το ΝΑΤΟ. Γι' αυτό πρέπει να θυμόμαστε ποιος είναι ο στόχος μας. Ο πρώτος στόχος πρέπει να είναι η ειρήνη και η συμφιλίωση στα Βαλκάνια. Με τα μέσα αυτού του κονδυλίου θέλουμε να υπηρετήσουμε αυτόν ακριβώς τον στόχο. Οι σωστές ε, γειτονικέ σχέσεις, συνεργασία και δικτύωση των χωρών και μεταξύ των διαφορετικών εθνοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος δωρητής στην περιοχή, αλλά ένα τεράστιο ποσοστό των ανθρώπων εκεί δεν το γνωρίζουν καν. Οι άνθρωποι της περιοχής όμως πρέπει να γνωρίζουν ποιος είναι αυτός που τους στηρίζει. Προφανώς ε, πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας για να ακουστούμε. Άλλες χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία, η Τουρκία, οι αραβικές χώρες ε, ήδη επενδύουν και, και εδώ και χρόνια. Όμως οι επενδύσεις αυτές ε, δεν έχουν τόσο καλούς στόχους όσο οι δικές μας. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να διαφημίζουμε την καλή δουλειά που κάνουμε. Τα στατιστικά στοιχεία μας λένε πως η οικονομία στις υποψήφιες χώρες αυτές αναπτύσσεται, όμως στην πραγματικότητα δεν βλέπουμε κάποια ουσιαστική βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Η ανάπτυξη δεν δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Οπότε ελήψη προοπτικών, πολλοί άνθρωποι από τις χώρες αυτές δεν βλέπουν καμία άλλη διέξοδο από τη μετανάστευση. Γι' αυτό είναι σημαντικό για εμάς το μέσο αυτό να μην εξαντληθεί στο να δίνει βοήθεια στις κεντρικές κυβερνήσεις, στις πρωτεύουσες, αλλά και στις υπόλοιπες περιφερειές. Και εκεί πέρα βέβαια, δεν παίζει κανένα ρόλο ε, ποιο κόμμα έχει την πλειοψηφία. Το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων πρέπει να βελτιωθεί και βεβαίως ε, χέρι-χέρι πηγαίνει η ευημερία με τη δημοκρατία. Η οικοδόμηση θεσμών, εκδημοκρατισμός, ε, δημιουργία κράτους δικαίου είναι η βασική μας στόχη. Και το κράτος δικαίου δεν είναι δώρο προς τον κύριο Γιούνκερ ή τον κύριο Τούσκ ή τον επίτροπο Χάν η τήρησή τους και η εφαρμογή τους από το χαμηλότερο μέχρι τα υψηλότερα επίπεδα της κοινωνίας είναι μια υποχρέωση και του κράτους και των πολιτών. Χωρίς το κράτος δικαίου δεν μπορεί ούτε να εγκριθεί ούτε να εφαρμοστεί σωστά το κοινοτικό δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει και την αξιοπιστία της ε, όταν ζητάει αυτές τις αξίες από τις υποψήφιες χώρες, ενώ ταυτόχρονα κάποια κράτη-μέλη δεν τις σέβονται. Γι' αυτό θα πρέπει να αποτελέσουμε το καλό παράδειγμα πρώτα εμείς αγαπητοί συνάδελφοι. Θεωρώ ότι έχουμε μια πολύ καλή έκθεση. Να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές και τους κοιοδησηγητές και είμαι σίγουρος ότι αύριο θα έχουμε μια ευρία πλειοψηφία για να κάνουμε το επόμενο βήμα και προς το συμφέρον των φίλων μας στα Δυτικά Βαλκάνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς κύριε Φλέκενστάιν και τώρα τον ρόλο έχει ο Επίτροπος, ο κύριος Χάν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Θα ήθελα να σε συγχαρώ, ιδίω στους δύο εισηγητέ για την εξαιρετική τους εργασία. Χαίρομαι πάρα πολύ, βλέποντα τη θέση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, βλέπω ότι υπάρχουν πολλά σημεία σύγκληση. Όχι μόνο, όσον αφορά τη νέα προγραμματική περίοδο, αλλά είναι αυτή η πρόταση χρηματοδότηση για τον νέο μηχανισμό προταξική βοηθεία 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την ασφάλεια και την ευμερία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται λοιπόν για ένα μηχανισμό που επιτρέπει στου εταίρου μα να ενισχύσουν του δημοκρατικού του θεσμού, να ενισχύσουν το δικαστικό σύστημα, να ενισχύσουν την οικονομία του και να έχουν ουσιαστικά πρότυπα ευρωπαϊκά για την προστασία των καταναλωτών αλλά και για το περιβάλλον. Όλα αυτά τα ωφέλη ουσιαστικά ωφελούν τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ε, τρίτες χώρες. Αυτή τη στιγμή θα έχουμε θεματικέ προτεραιότητες στο πλαίσιο του ΙΠΑΤΡΙΑ και όχι τόσο πολύ χορηγήσει ανά χώρα. Θα έχουμε επίση μια προσέγγιση που θα βασίζεται σε πραγματικέ επιδόσεις. Είναι πολύ σημαντικό να πετύχουμε την απαραίτητη ισορροπία ανάμεσα στου στους στόχου, προκειμένου να μπορούν οι χώρε εταίροι να καταρτήσουν στου προ... σωστούς αλλά από την άλλη θα πρέπει να έχουμε και τι σωστέ επιδόσει από τι χώρε αυτέ, ώστε να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε αυτές που πετυχαίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Επίσης, είναι σημαντικό να υπάρχει η καλύτερη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο πλαίσιο της θεσμικής ισορροπίας της συνθήκες θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να προωθηθεί περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό θα το εξετάσουμε περισσότερο στα πλαίσια του μερούς διαλόγου που ελπίζουμε να ξεκινήσει στο Μότρο δυνατό. Ένα ζήτημα το οποίο θέλω να θέσω είναι το να καταφέρουμε να τηρήσουμε την ε, ισορροπία δράση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Χρειάζεται συνέπεια ανάμεσα στην πολιτική διεύρυνση και την εξωτερική πολιτική. Αυτή τη στιγμή, μέσω του μηχανισμού αυτοπροταξιακή βοήθεια, θέλουμε ουσιαστικά να καταφέρουμε να προωθήσουμε αυτή την ε, ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική. Μέσω της πολιτικής αυτής ουσιαστικά προωθούμε περισσότερο την εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν προτείνετε εσείς έναν συγκεκριμένο μηχανισμό στην έκθεση αυτή θα πρέπει να ξεχνάτε ότι αποτελεί ουσιαστικά μία επικάλυψη σε σχέση με ζητήματα τα οποία έχουμε ήδη εμείς προτείνει. Όσον αφορά τώρα Του συντελεστέ Gini και αυτοί θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να έχουμε καλύτερη συνέπεια και συνεκτικότητα όταν αντιμετωπίζουμε του εξωτερικού μα εταίρου. Και στόχος σας προφανώς δεν είναι να υπονομεύσετε εσείς τους στόχους αυτούς, αλλά καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν διαφορετικές διαπραγματεύσεις όσον αφορά το ΙΠΑ και το ΛΥΚΙ και θα πρέπει να καταφέρουμε να έχουμε τελικά κοινούς κανόνες. Σας ευχαριστώ πολύ για την έκθεση σας αυτή. Eh, Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Μπορέλη εκ μέρους της Επιτροπής ε, Διεθνούς Εμπορίου. Αλλά δεν το βλέπω στην αίθουσα, οπότε περνάμε στην εκπρόσωπο της Επιτροπής Προϋπολογισμών, την κυρία Ιβάνα Μάλετιτς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, Καλωσορίζω και τον Επίτροπο Χάν που είπε για ποιου τομεί είναι απαραίτητο ο μηχανισμό προδεξιακή βοήθεια. Τώρα έχουμε νέε προκλήσει, όχι μόνο στη, των χωρών μελών, αλλά και των υποψήφιων για ένταξη χωρών. Ε, τα θέματα του περιβάλλοντο, τη ενεργειακή απόδοση, μετανάστευση είναι νέε προκλήσει και για τι υποψήφιε για ένταξη χώρε. Θα πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε στον προπολογισμό του μηχανισμού αυτού αρκετά κονδύλια και για τι νέε προκλήσει. Και χρειάζεται και στρατηγικό ε, σχεδιασμό προορατικός. Δεν συμφωνώ με την κατανομή των κονδυλίων μόνο με βάση θεματικές προτεραιότητες και όχι ανάλογα με τις χώρες δικαιούχους. Είναι σημαντικό να έχουμε ενδεικτικά ποσά αναχώρα, υποψήφια για ένταξη χώρα και όχι μόνο θεματική κατανομή των κονδυλίων, γιατί στις χώρες που δεν υπάρχουν αρκετά προγράμματα ή δεν υπάρχουν αρκετές ικανότητες, δεν υπάρχουν αρκετές προτάσεις, θα πρέπει αυτές τις χώρες να βοηθήσουμε με τεχνική αρρωγή, αλλά και με διοικητική ενίσχυση των αντιπροσωπιών μας, ώστε να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα κονδύλια αυτά και όχι μόνο να ανταγωνίζονται μεταξύ τους ε, και οι καλύτεροι να προχωρούν ενώ οι λιγότερο καλοί και ανεπτυγμένοι να μένουν πίσω. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, για ένα λεπτό κύριο Τζέλερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επιτροπή πολιτική αυτή της πρωταξιακής βοήθειας είναι από τις πιο επιτυχημένες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πολλά κράτη-μέλη κατάφεραν έτσι να βρουν τον δρόμο τους ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως οι άνθρωποι στις χώρες αυτές βλέπουν το, μέλος τους, το μέλλον τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως η διαδικασία στις περισσότερες από αυτές τις χώρες πηγαίνει πάρα πολύ αργά ή στην περίπτωση της Τουρκίας έχουμε και οπισθοδρόμηση, γιατί επικεντρώνεται κυρίως στην κυβέρνηση, ειδικά για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και τους ανθρώπους εκεί. Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωση είναι ακριβώς κάτι το οποίο βοηθάει από κάτω, ε, προς τα πάνω βοηθάει την βάση. Και έχουμε ακριβώς ε, την συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και ε, της ε, τοπικής αυτοδιοίκησης ε, στις χώρες αυτές, κάτι το οποίο θα καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ορατή στις χώρες αυτές, κάτι το οποίο δεν γίνεται αυτή τη στιγμή, τα είπε ο κύριος Φλέκενστάιν. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα της συνεργασίας και της επέκτασης αυτού του μέσου. Ελπίζω λοιπόν να το εκμεταλλευτούν και να το αξιοποιήσουν πλήρως. Σας ευχαριστώ κύριε Τσέλερ από την Επιτροπή Ελευθεριών και Εσωτερικών, η κυρία Βαλέρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να επαναλάβω πως το μέσο πρωτεξιακής βοήθειας 3 είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καμιά φορά πηγαίνουν σε λάθος κατεύθυνση τα κονδύλια αυτά. Καταλήγουν παραδείγματος χάρη σε τεθωρακισμένα οχήματα ή ε, οχήματα για περιπολίες στην Τουρκία για να εμποδίσουν την μετανάστευση. Ε, υποτίθεται ότι δεν πάνε σε εξοπλισμούς. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον ε, το ότι μπορούν να στηρίξουν τέτοιες δυνατότητες. Θα μπορούσαν δηλαδή να χρησιμοποιηθούν για την αγορά τέτοιων οχημάτων από την Τουρκία που μετά τα χρησιμοποιεί στις συγκρούσεις με τους γειτονές της. θα πρέπει να πάνε στη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, ε, λιγότερες διακρίσεις. Επίσης σημαντικό είναι τα μέσα αυτά να μπορούν ε, να ανασταλούν όταν μια χώρα δεν σέβεται τις ευρωπαϊκές αξίες και να πάνε στην κοινωνία των πολιτών που βοηθάει στην εφαρμογή των δικαιωμάτων αυτών. Χρειάζεται λοιπόν καλύτερος έλεγχος και περισσότεροι όροι. Σας ευχαριστούμε κυρία Βαλέρο. Τώρα από το ΕΛΚΟ, ο κύριος Πρέτα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που συνεχίζουμε τη συζήτηση που ξεκινήσαμε πριν από λίγο. Χαίρομαι πάρα πολύ που η δική μου χώρα γλίτωσε από την προσπάθεια αυτή να μπουν όλα μέσα σε αυτό το ενιαίο μέσο. Ο κύριος Παντσέρη προσπαθούσε να βάλει ακόμα και το ΙΠΑ στο Μηχανισμό Γειτονίας Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους Ιγνάθιο και Κνούτ για την εξαιρετική τους εργασία. Τα προταξιακά κονδύλια αποτελούν μακροπρόθεσμη επένδυση για το ευρωπαϊκό μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων και είναι πολύ σημαντικό η χρηματοδότηση αυτή να επανασυγκεντρωθεί προκειμένου να έχουμε μία πρόοδο ξεκάθαρη και μία αναστρέψιμη για τομεί κλειδιά βάσει των κριτηρίων τη Κοπενχάγη. Είμαι υπέρ τη γενικότερη φιλοσοφία τη έκθεση αυτή και τη ενίσχυση ερεσιμότητα όσον αφορά την οικονομική συνδρομή. Η βασική αλλαγή όσον αφορά το ΙΠΑ 3 μέσω τη αρχή τη δίκαιη κατανομή θα αποτελέσει πραγματικά κίνητρο, θεωρώ, για μεγαλύτερη ευθύνη, λογοδοσία και πιο σοβαρή στάση από τι εμπλεκόμενε χώρε. Να ευχαριστήσω επίση του ηγητέ που έλαβαν υπόψη τροπολογίε μου για δύο σημεία. Πρώτον, να έχουμε μια καλύτερη συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών και να έχουμε την υποστήριξη στι δικαιούχε χώρε τη αποϊδρυματοποίηση των παιδιών. Σα ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρέντα. Εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών τώρα, ο Τονίνο Πίτσουλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Η χρηματοδότηση του μηχανισμού Προταξιακής βοήθειας είναι μακροπρόθεσμες επενδύσεις στο ε, ευρωπαϊκό μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων. Βέβαια, το μέλλον αυτό γίνεται όλο και πιο αβέβαιο, δεδομένου του πολιτικού κλίματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των προκλήσεων που αντιμετωπίζει και των επερχόμενων εκλογών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα πρέπει πάντως να δώσουμε ευκαιρία στα Δυτικά Βαλκάνια να εκπληρώσουν τα κριτήρια και να προετοιμαστούν για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Μαυροβούνιο έχει προχωρήσει πολύ στο, στις πρωτεξιακές διαπραγματεύσεις και η Βόρεια Μακεδονία έχει κάνει μεγάλο δρόμο και αξίζει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις διαπραγματεύσει και η Αλβανία το ίδιο. Θα πρέπει λοιπόν με τα μέσα αυτά να τονωθεί η ανάπτυξη στις χώρες αυτές, η πρόωθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης να στηρίξουμε τη δημιουργία ικανοτήτων και να επιτρέψουμε την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και των υποψηφίων χωρών. Επίσης, ε, λυπούμαστε που κάποιες ε, προτάσεις μας δεν έγιναν δεκτές. Παρόλα αυτά, συγχαίρω τους συνεισηγητές και σας συστήνω την υπερψήφιση της έκθεσης. Σας ευχαριστούμε κύριε Πίτσουλα. Εκ μέρους του ΙΣΙΑΡ τώρα, ο κύριος Δεμεσμάκερ έχει το λόγο. συχνά εδώ πέρα ζητάμε η Κομισιόν να δει τον τρόπο με τον οποίο στηρίζουμε την ε, Τουρκία. Δεν έχουμε ενισχύσει τη δημοκρατία, το αντίθετο μάλλον. Έχουμε λοιπόν πρωταξιακά προγράμματα τα οποία έχουν εδώ πέρα ενδιάμεσες αξιολογήσεις με μια καλύτερη αιρεσιμότητα. Ελπίζουμε λοιπόν πραγματικά να πάει το μήνυμα στον κύριο Ερντογάν. Το μόνο μάθημα το οποίο μπορούμε να αντλήσουμε από τις εμπειρίες του παρελθόντος είναι ότι δεν είναι ανάγκη να δίνουμε το βάρος σε μελλοντική διεύρυνση αλλά σε καλή γειτονία. Το προενταξιακό μέσο λοιπόν δεν είναι εδώ πέρα το καταλληλότερο μέσο. Αυτά τα οποία περιέχονται, δηλαδή η στήριξη του κράτου, δικαιώτα, θεμελιώδη δικαιώματα, η ορθή χρηστή διοίκηση κτλ. είναι επίση να χρηματοδοτηθούν από τα άλλα εξωτερικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστούμε κύριε Ντεμέ Μάκερ. Τώρα εξ ονόματο της Άλντε τον λόγο έχει ο κύριο Κιτσούκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Από το 2007 το μέσο πενταξιακής βοηθείας είναι το κύριο χρηματοδοτικό μέσο το οποίο στηρίζει τις υποψήφιες χώρες ε, των ε, Βαλκανίων ε, και της του Έχουμε λοιπόν μια στρατηγική εστίαση στα έγγραφα αυτά ανά χώρα που εστιάζουν στον στρατηγικό σχεδιασμό. Καλωσορίζω λοιπόν εδώ πέρα την πρόταση της Κομισιόν για ένα μέσο πρωτεξιακής βοηθείας υπαριθμών 3. Ε, Βεβαίω ε, δεν έχει οδηγήσει σε τεράστιες επιτυχίες τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό ακριβώς χαιρετίζω το ότι εστιάζει πλέον στο κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την μετανάστευση τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, το ευρωπαϊκό και εκτιμένο και τις, ε, καλές, ε, και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Συγκεκριμένα λοιπόν ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να γίνει όχι μόνο σε συνδυασμό με την στρατηγική